Hello everyone, please. Καλησπέρα σε όλους σας, παρακαλώ καθίστε. Ε, ήταν ε, πολύ φορτισμένη συγκινησιακά αυτή η μέρα, πραγματικά ιστορική ημέρα σήμερα ε, και ερχόμαστε από μια ψηφοφορία η οποία αλλάζει το Κοινοβούλιο, αλλάζει την ίδια την Ευρώπη έτσι όπως την ξέραμε και βεβαίως τώρα θα πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον γιατί είναι το μόνο που μπορούμε πλέον να κάνουμε. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην συνεδρίαση αυτή, στη συνάντηση αυτή. Είναι η πρώτη, ε, η πρώτη συνάντηση του πάνελ ΣΤΟΑ για αυτήν την περίοδο. Έλεγα ότι είναι φορτισμένη συγκινησιακά η μέρα αυτή. Ωστόσο τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε για τα πιο ωραία πράγματα τα οποία περιμένουν και έρχονται μπροστά μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ ε, στη διάρκεια της συζήτησης ε, θα υπάρχει και διάδραση με το ε, Twitter γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να τα κάνουμε όλα πολύ σωστά αυτή τη φορά. Θέλουμε τώρα να συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο για τις νέες τεχνολογίες, καθώς επίσης και τις αναδυόμενες ε, επιστήμες. Ε, ξέρετε ότι αυτή η Επιτροπή λειτουργεί εδώ και 25 χρόνια ε, και ασχολείται με ένα σωρό τομείς ε, όπως εφηή σπόροι, ε, τεχνητή νοημοσύνη, ενέργεια, γεωργία κλπ. Και βεβαίως έχουμε ένα σύστημα εμπλεκομένων επιστημόνων κλπ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, κυρία Φεστάγκερ γιατί αποδέχτηκε την ε, πρότασή μας. Ε, είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαστε εδώ μαζί σας, που είμαι δίπλα σας. Είστε μια δυναμική πολιτικός, ε, είσαστε μια δυνατή γυναίκα που μπορεί να αφήσει και θα αφήσει το αποτύπωμά της στην Ευρώπη. θα, όπως το επιθυμούσατε άλλωστε και εκφράσατε αυτή την επιθυμία, θα κάνουμε μια συζήτηση ε, και θα έχουμε και fireside chat με τον Άντων και τον Ανδρέα Ρέντα έτσι ώστε να συζητήσουμε για όλες τις ψηφιακές προκλήσεις. Νομίζω ότι όλοι με ενθουσιασμό περιμένουμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά, γιατί ε, η παγκοσμιοποίηση βεβαίως μπορεί να ενέχει κάποιες δυσκολίες, αλλά αποτελεί και μεγάλη πρόκληση. Είναι προκλήσεις αυτές ε, οι τεχνολογίες της αλυσίδας στοιχειών, blockchain και άλλες. Επομένως, ε, είναι γεγονός ότι υπάρχει και το παράδοξο ότι παρότι αυτές οι τεχνολογίες δεν γνωρίζουν σύνορα, πρέπει να καθορίσουμε και κάποιους κανόνες, όπως α πούμε είναι η αμοιβαιότητα, η προστασία της ιδιωτικότητας, η προστασία της δημοκρατίας, η προστασία της ε, κυριαρχίας, αλλά χωρίς προστατευτισμό. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην καινοτομία και όλα αυτά, ο συνδυασμός δηλαδή όλων αυτών δεν είναι πάρα πολύ εύκολος. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε ε, τουλάχιστον αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα αρκετά καλά, να προστατέψουμε την ιδιωτικότητα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η νομοθεσία βέβαια για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν ε, για την ε, θέση σας. Εσείς ε, έχετε περάσει από πολλές ε, θέσεις από το Κοινοβούλιο της Δανίας, είχατε υπουργικό ε, θόκο, επίσης έχετε μεγάλη εμπειρία, άρα είστε πραγματικά ο άνθρωπος που χρειάζεται για την θέση αυτή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις ηθικές, οικονομικές, δεοντολογικές κλπ. Και θα σας δώσω τον λόγο έτσι ώστε να μας κάνετε μία πρώτη ε, εισαγωγή. Uh, Είσαστε πολύ ευγενικοί, αλλά νομίζω ότι αυτά συμβαίνουν σε μέρες τέτοιες φορτισμένες. Ε, Ήταν πολύ συγκινητική ε, μέρα και ξέρω ότι Ε, δεν μπορώ να τα αλλάξω αυτά, ούτε δεν μπορώ να γυρίσω πίσω το χρόνο. Θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει πριν από μισή ώρα. Ε, λίγο μετά τις 7 θα πρέπει να σας εγκαταλείψω δυστυχώς. Ε, θα κάνω λοιπόν μια σύντομη πρώτη παρέμβαση και μετά ελπίζω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, ε, διότι είναι δύσκολα τα θέματα αυτά και αν δεν τα ε, συζητήσουμε δεν θα τα κάνουμε σωστά από την αρχή. Δεν ε, υπάρχει ε, κάποιο κεντρικό μυαλό που να μπορεί να τα κάνει αυτά, διότι η υπόσχεση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι θα έχουμε νέο εργαλείο για να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας. Ε, υγεία για όλους και για ανθρώπους που πάσχουν από ασθένειες τις οποίες άλλοι δεν έχουν καν ακούσει έλεγχος της κυκλοφορίας, καταπολέμηση της αλλαγή του κλίματος, διότι θα γνωρίζουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους μας και να πραγματοποιήσουμε την κυκλική οικονομία. Το θέμα είναι όμως ότι για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε την τεχνολογία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η εμπιστοσύνη μειώνεται. Και όχι λόγω της τεχνητής νοημοσύνης αυτής καθ' αυτής, ε, δεν νομίζω, αλλά επειδή ε, δημοσιεύονται φωτογραφίες που δεν θα έπρεπε να δημοσιεύονται, περίεργα email, απειλές και ένα σωρό περίεργα πράγματα που συμβαίνουν. Για να οικοδομήσουμε λοιπόν εμπιστοσύνη πρέπει να συζητάμε και πρέπει να δείξουμε στους ανθρώπους ότι όταν είναι επικίνδυνα τα πράγματα θα είμαστε στο πλευρό τους. Έχουμε λοιπόν αυτή την διτή προσέγγιση ένα οικοσύστημα εμπιστοσύνης και ένα οικοσύστημα αριστείας. Το οικοσύστημα αριστείας ε, οικοδομείται χρησιμοποιώντας σωστά τους σπόρους διαθέτοντας τους ε, απαραίτητους σπόρους ε, για να υπάρχουν δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και για να προσελκύσουμε ταλέντα, να προσελκύσουμε καλά μυαλά. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι έχουμε τεράστιο χάσμα όσον αφορά ε, τα δύο φύλλα, ε, όταν βλέπουμε ποιοι ασχολούνται με αυτές τις τεχνολογίες. Όσον αφορά την εμπιστοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται παντού. Ήδη βρίσκεται στα κινητά μας τηλέφωνα, μας βοηθάει στη μετάφραση, ε, έλεγχο της φωνής, ε, οι λίστες τραγουδιών ε, στους υπολογιστές και ακόμη και αν η υπηρεσία μουσική που χρησιμοποιώ μου δώσει τραγούδια που δεν μου αρέσουν, θα βρω άλλα. Δεν πειράζει, αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Αλλά αν η τεχνητή νοημοσύνη με βοηθεί, βοηθάει το γιατρό μου να καταλάβει τι είδου καρκίνο έχω, ε, τότε είναι τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Όταν ε, λοιπόν είναι θέμα ζωή και θανάτου, ε, θα πρέπει να είμαστε ε, πολύ πιο αυστηροί για να είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί, μπορούμε να την εμπιστευτούμε, να όσον αφορά την ε, ποιότητα, τα δεδομένα, ε, το πόσο εύκολο είναι να ε, εξηγηθεί στους πολίτες. Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους τεχνολογίες. Και υπάρχει μια τρίτη διάσταση που έχει να κάνει με τις ευαίσθητες τεχνολογίες. Σε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, ματιών, φωνής, περπατήματος, του βηματισμού μας, των κινήσεων του σώματός μας. Ε, εδώ υπάρχει ο κίνδυνος ε, υπονόμαυσης ε, των θεμελιωτών δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε να διαμαρτύρεται κανείς μαζί με άλλους ανθρώπους και έχουμε ανοιχτή ελεύθερη κοινωνία και γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να γνωρίζουμε τι κάνουμε όλοι και να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτά. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα με τη σημερινή πρωτοβουλία. Χαίρομαι που ε, ε, είμαστε εμείς εδώ οι τέσσερις και ότι είναι τόσο γεμάτη αίθουσα, διότι είναι μια συζήτηση που αφορά όλους. Στις 19 Φεβρουαρίου ε, θα ξεκινήσουμε τη στρατηγική με βάση μια λευκή βίβλο και έτσι θα ξεκινήσει η συζήτηση και θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να επανέλθουμε στο θέμα. Σας ευχαριστώ. Ήταν αποτελεσματική και σύντομη παρέμβαση. Έχουμε ερωτήσει. Παρακαλώ τους συναδέλφους να ξεκινήσουν. Ποιο θέλει να μιλήσει. Πέτρα, Τιέμο. Πέντε ερωτήσει θα ακούσουμε και μετά θα κάνουμε δεύτερο γύρο απαντήσεων. Μία Πέτρα. Ευχαριστώ, Εύα θα πάω κατευθείαν στην ερώτηση. Περιμένουμε τη λευκή βίβλο. Συζητείτε τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται λόγος, θα υπάρξει κανονισμός. Κάποιες εταιρείε φοβούνται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεσπίσει νομοθεσία, φοβούνται εταιρείε την νομοθεσία και τον κανονισμό. Θα υπάρχουν κανόνες σχετικά με το πώς, ποιος κωδικοποιεί τα βασικά στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης. Θα ωφεληθούν και εταιρείε όταν ξέρουν περί αυτών. Όταν χαθεί ο, αυτός που κωδικοποιεί το σύστημα, πρέπει κάπου να αποθηκεύεται το κωδικοποιημένη βάση. και να πρέπει να ξέρουμε να υπάρχει και η χνηλασιμότητα του κωδικά που παράγεται, πώς έχει παραχθεί, από πού προέρχεται και όλα αυτά. Δύσκολη ερώτηση. Και έξοχη. Ο κύριος Σαλίμπα, ε, Πατρίτσια, η Πατρίτσια Τόγια. Ευχαριστώ, θα μιλήσω Ιταλικά, κύριε Βεστάγκερ. Ήθελα πάνω απ' όλα να συγχαρώ για την ε, προσπάθεια που κάνατε. Ήδη και στην Ήτρε έχει τεθεί ε, αυτός ο στόχος και τα καθήκοντα εκτελείται. Ποια είναι η εμπειρία μου. Οι επιχειρήσεις περιμένουν έναν κανονισμό, μια ρύθμιση. Εγώ δεν πιστεύω ότι φοβούνται. Ίσως υπερβολικό, ε, υπερβολική νομοθεσία φεύγονται, αλλά θέλουν κάτι για τις διάφορες πτυχές που εμπλέκονται. Το δεύτερο που αναφέρατε σε κάποια παρέμβαση και είναι κρισίμου σημασίας είναι το θέμα όχι τη ιδιοκτησία των δεδομένων, αλλά η χρήση των δεδομένων. Χρήση προποθέτει βέβαια και ιδιοκτησία. Τα ε, open assets, ε, η έρευνα, έγινε αρχή ευρωπαϊκή φορέας για την έρευνα. Είναι σωστή προσέγγιση. Ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι σε καλύτερη θέση να παίρνει αυτά τα στοιχεία και να τα χρησιμοποιεί τα δεδομένα πιο σωστά. Όπως τα κοινά αγαθά που συζητήσαμε. Η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή. Ε, τέλος, πρίμα την, τις κατευθυντές γραμμές, μιλήσαμε στην Ευρώπη για αδελογικές αρχές. Από τους stakeholders νιώθω ότι επικρατεί κάποια βεβαιότητα. Δεν λέω υποτίμηση, αισθάνονται ότι υπάρχει κάποια υποτίμηση. Σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω ότι πιστεύουν και αυτοί ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι κάτι ε, ισχυρό, ισχυρό σημείο. Περιμένουμε πολλά από εσά. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη, αλλά περιμένουμε από εσά και μεγάλα αποτελέσματα. Ε, μου, όσο πιο σύντομα μπορείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που ήρθατε ξανά. Ήσασταν παρούσα και συζητήσει στην Νομική Επιτροπή. Αυτό δείχνει πώς αφοσιωμένοι είσαστε να διατηρήσετε καλό διάλογο με το Κοινοβούλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Όλοι περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει τα μέτρα στις πρώτες 100 μέρες για την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρουμε ότι θα είναι μια λευκή βίβλος. Έχω δύο ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 αναφέρει ότι θα πρέπει να κατατήσουμε ένα οικοσύστημα εμπιστοσύνης. Συμφωνώ απόλυτα με αυτή την προσέγγιση και βλέπουμε ότι κάποια κράτη-μέλη ήδη κινούνται προς τα μπρος. Στη Γερμανία υπάρχει μια επιτροπή για τη δεντολογία των δεδομένων, έχει κάνει κάποια σύσταση, η Δανία ήδη σκέφτεται το να θεσπίσει μια σφραγίδα διοντολογική για τα δεδομένα, ήδη εξετάζουν τα διάφορα κράτη-μέλη τα μέτρα τους και προσπαθούν να εφαρμόσουν πολύτιμες συστάσεις του επιστημονικού κόσμου. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα υπάρξει ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη που θα επιτρέπει αρκετά περιθώρια για να δημιουργηθούν οικοσυστήματα, αλλά να είναι ακόμα αποτελεσματικό. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Η καινοτομία είναι σημαντικότατη για την ε, οικονομία των δεδομένων και το ίντερνετ των πραγμάτων και τη βιομηχανία, την καινούρια που δημιουργείται στην Ευρώπη. Αν μιλάμε για αξιόπιστη όμως ε, τεχνητή νοημοσύνη, ποια, τι συνεπάγεται ότι η προσέγγιση μας στην τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Κατά την άποψή μου αυτό είναι μόνο εφικτό αν το ρυθμιστικό μας πλαίσιο για τεχνητή νοημοσύνη εδράζεται στερεά στην αρχή της πρόληψης, η προστασία των δεδομένων αναφέρεται στο GDPR, και χρειάζεται μέτρα διαφύλαξη για τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπω και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ίσως μπορείτε να λήξετε φως σε αυτό, πώς μπορείτε να πετύχετε την απαιτούμενη α, ισορροπία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, ξέρετε ότι εγώ έρχομαι από την πολιτική ομάδα ΡΙΝΙΟΥ, επομένως δεν είναι μυστικό ότι εδώ και αρκετό χρόνο εμείς προσπαθούμε να ε, έχουμε ένα ε, κοινό έγγραφο όσον αφορά την, ε, το έγγραφο θέσης για την τεχνική νοημοσύνη. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι η ίδια η άσκηση της τεχνικής νοημοσύνης θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο έγγραφο θέσης. Βεβαίω έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες έτσι ώστε ε, να βρούμε αυτή την κοινή συνισταμένη ανάμεσα στην ανάγκη ανάπτυξη, στην ανάγκη προστασίας δεδομένων κλπ. Και φυσικά και την ανάγκη να βρούμε αυτήν την χρυσή γραμμή ανάμεσα στην προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων από τη μία και την ανάπτυξη αξίας από την άλλη μέσω τη χρήση των δεδομένων. Πού πιστεύετε ότι θα καθίσει τελικά ο Κέρσορα όσον αφορά αυτά τα ε, δύο αντιτιθέμενα σε μια πρώτη φάση και εκ πρώτης όψεως στοιχεία. Επίσης, ε, ε, συζήτηση γίνεται για πολλούς μήνες για το ίδιο θέμα και το ερώτημα το οποίο προκύπτει από την βιομηχανία είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα sandbox βάσει του οποίου θα δημιουργηθεί ή τέλος πάντων θα παρακινήσουμε την δημιουργία ενός ορθού πλαισίου το οποίο θα λειτουργήσει εντός ασφαλούς περιβάλλοντος. και η βιομηχανία χρειάζεται ταλέντα έτσι ώστε να αναπτύξει τις τεχνολογίες αλλά και οι δημόσιες, δημόσιες αρχές από τη δική τους πλευρά χρειάζονται αυτό το ταλέντο έτσι ώστε να ελέγξουν, να ελέγχουν ε, και να αξιολογούν αυτήν την ε, τεχνολογία, την εξελισσόμενη τεχνολογία. Θα ήθελα τις απόψεις σας γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κριστόφ και μετά θα απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ Εύα που οργάνωσες ε, αυτήν την ε, συνάντηση. Κυρία Επίτροπε, ποια θα είναι η προσέγγιση της Κομισιόν όσον αφορά την διευκόλυνση πρόσβασης των δεδομένων. Ε, προτείνεται ή θα προτείνεται κάποια αναθεώρηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων GDPR ε, Μεγάλη ανησυχία έχει προκύψει βάσει ε, λόγω του άρθρου 5 ε, του κανονισμού που αφορά την συλλογή και χρήση των δεδομένων. Πώς προτίθεστε να βρείτε την χρυσή γραμμή ανάμεσα το να δημιουργήσετε ένα ασφαλές πλαίσιο το οποίο να ε, εγγυάται την προστασία των δεδομένων από τη μία και τις ανάγκες ανάπτυξης και δεδομένων που έχουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από την άλλη. Επίσης, ε, προτίθεστε για τομείς όπως η υγεία να έχετε πιο αυστηρή τομεακή προσέγγιση. Επίσης, ποια είναι η θέση σας όσον αφορά την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Πολύ απλέ ερωτήσει, λέει η Πρόεδρος, να έχουμε τις πρώτες απαντήσει από την κυρία Επίτροπο. Θα ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση όσον αφορά την αναγνώριση χαρακτηριστικών προσώπου και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά του σώματος για ταυτοποίηση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι αν δεν είμαστε υπάρχει ο κίνδυνος η πρόχειρη εφαρμογή να υπονομεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα στα συντάγματά μας, ε, στη συνθήκη και λοιπά. Εγώ δεν θα απέκλεια ποτέ ότι οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να είναι ασφαλείς και χρήσιμες, αλλά νομίζω ότι είναι ε, σημαντικό να έχουμε, απαραίτητο, να έχουμε επαρκή χρόνο ώστε να το διασφαλίσουμε αυτό. Υπάρχουν τεχνολογίες ευαίσθητες, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να ε, υπονομεύσουν ε, ακριβώς ε, τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις κοινωνίες μας όσον αφορά την ηθική, τη διεντολογία. Για μένα το πρώτο βήμα είναι αυτό που σχετίζεται με τον κίνδυνο. Σε κάθε τομέα υπάρχουν πράγματα τελείως ακίνδυνα ή τόσο όχι πολύ επικίνδυνα και πράγματα ζωτικής σημασίας για την ευημερία, πιθανότατα και θέματα ζωής ή θανάτου. Ε, και σε οποιονδήποτε τομέα θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν είναι τεχνολογία υψηλού κινδύνου, να υπάρχει πλαίσιο που να τη ρυθμίζει, να υπάρχει διακυβέρνηση και σωστή επιβολή των κανόνων. Και εγώ θα προτιμούσα να έχω απλά πράγματα με ε, ε, τεχνολογίες υψηλού κινδύνου παρά να έχω ε, ένα πολύπλοκο πλαίσιο ε, που να μην μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα. Να έχουμε δηλαδή απλούς κανόνες για τις τεχνολογίες αυτές. Όσον αφορά τα δεδομένα, ε, για μένα σημαντικό είναι να εφαρμοστεί πλήρως ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων, όχι να τον αναθεωρήσουμε. Ε, οργανισμός προστασίας, οι φορείς προστασίας δεδομένων ακόμη μαθαίνουν, το κάνουν αυτό κάθε μέρα. Νομίζω όμως ότι έχουμε ακόμα πράγματα να κάνουμε για να νιώσουν οι πολίτες ότι έχουν τον έλεγχο με ε, τον ε, κανονισμό για τα δεδομένα ε, έχουμε καλά δικαιώματα, έχουμε τα σωστά δικαιώματα, αλλά θα πρέπει να μπορεί να τα ασκήσει κανείς. Από την άλλη, υπάρχουν τόσα πολλά άλλα δεδομένα που δεν είναι προσωπικά, δεδομένα που καλύπτονται από τον κανονισμό. Σκεφτείτε το διαδίκτυο των πραγμάτων, το Internet of Things. Θα είναι τεράστιος ο όγκος δεδομένων που θα παράγονται. Ε, υπάρχουν ε, δεδομένα επιχειρήσεων, υπάρχουν ε, δεδομένα μηχανών και πολλές επιχειρήσεις λένε ότι, ε, μου λένε ότι τα δεδομένα αυτά είναι χρυσό. Ε, αν είναι χρυσό, δεν θέλω να τα μοιραστώ με κανέναν. Εάν όμω δεν τα μοιραστείτε τότε ε, χάνεται και η αξία του. Ε, πολλοί κόσμος ε, δεν γνωρίζει πώ πρέπει να τα χρησιμοποιήσει αυτά. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει να, βοηθήσουν, να χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα που ήδη έχουν στα χέρια του για να αναπτύξουν τι επιχειρήσει του. Ε, πρόσφατα άκουσα για μια επιχείρηση που ε, μπορεί να επιθεωρεί συστήματα διαχείρισης ε, υδάτων ε, σε όλον τον πλανήτη επειδή έχουν έλεγχο των σχετικών δεδομένων. Όσον αφορά τα ταλέντα, τα μυαλά, πώς θα τα βρούμε. Αυτό είναι θέμα ε, εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, διαβίου μάθησης. Εκπαίδευση λοιπόν ε, είναι όμως ε, κεντρικής σημασίας ε, μέτρο αυτό, διότι αν δεν έχουμε τις απαραίτητες δεξιότητες ε, δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα αυτά, ούτε θα είμαστε ελκυστικοί για άλλους ανθρώπους ε, που να έχουν τις δεξιότητες αυτές. Ε, και Ε, αυτό δυσκολεύει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι εμείς έχουμε όλες τις προθέσεις, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν τα εργαλεία για να πραγματοποιήσουν τους στόχους. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, πρέπει να καλέσουμε, να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους δίνονται. Και οι άνθρωποι, ιδιαίτερα της δικής μου γενιάς, θα πρέπει να τους σπρώξουμε για να μάθουν περισσότερα, να γίνουν πιο φιλόδοξοι για να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και σε αυτούς τους τομείς. Ε, το θέμα των, ε, του sandbox, ε, του ε, χώρου ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, ε, ε, διότι θα πρέπει να ελέγχουμε τις νέες τεχνολογίες πριν τις απελευθερώσουμε, πριν, τις, πριν κυκλοφορήσουν γενικά, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για πιο επικίνδυνες τεχνολογίες και πού θα πρέπει να βάλουμε τον κέρσορα ανάμεσα στην έρευνα και ανάπτυξη, την ανάπτυξη και καινοτομία και τις αξίες μας. Είναι ε, σημαντικό να είμαστε φιλόδοξοι και να θέλουμε να πετύχουμε και τα δύο και να μην τα βλέπουμε αυτά ω πράγματα αντίθετα, διότι δεν νομίζω ότι όλε οι καινοτομίε είναι καλέ καινοτομίε. Ε, αν ε, κάποιος κακός σε ταινία James Bond ε, εφεύρει ένα νέο όπλο, αυτό δεν είναι καλό. Το έχουμε δει αυτό χιλιάδες φορές. Υπάρχουν καινοτομίες όπου λέμε όχι ευχαριστώ οι καινοτομίε που θέλουμε είναι οι καινοτομίε που είναι ε, ε, βασισμένες σε μια ε, σταθερή βάση φιλοδοξιών και επιχειρηματικού, επιχειρηματικής νοοτροπίας όπου νιώθουμε ότι έχει αναπτυχθεί με το σωστό τρόπο. Και έτσι φτάνω στο θέμα της εμπιστοσύνης και των μέτρων προφύλαξης. Το θέμα αυτό δεν είναι νέο στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, το κάνουμε αυτό εδώ και δεκαετίες. Πολύ συχνά σκέφτομαι τη γεωργία. Πολλοί γεωργοί είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά ε, την χρήση φυτοφαρμάκων ε, και μεταχειρίζονται καλά τα ζώα τους. Ε, υπάρχει όμως μια μικρή μειονότητα πιθανότατα που δεν προσέχει όσον αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων και δεν ε, μεταχειρίζεται καλά τα ζώα. Επειδή όμως δεν, δεν θέλουμε να ρισκάρουμε το, ούτε το θέμα των ε, πόσιμων υδάτων μας, ούτε το θέμα της ε, ευημερία των ζώων και γι' αυτό νομοθετούμε. Δεν είναι λοιπόν νέο ότι στην Ευρώπη λέμε είναι δημοκρατία, οι πολίτες έχουν εκπροσώπους ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τρομάξουμε τους πολίτες να πούμε ότι είναι καινοτομία, τα πράγματα προχωράνε γρήγορα και γι' αυτό να μην κάνουμε τα θεμελιώδη πράγματα, ώστε οι πολίτες να έχουν και τα δύο, να διασφαλίσουμε και τι θεμελιώδεις αξίες μας και να δώσουμε τη δυνατότητα για καινοτομία. Διότι αυτό με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. για τις επιχειρήσεις ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουν τα απαραίτητα στοιχεία και να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μια σφραγίδα ε, δεοντολογίας όσον αφορά τα δεδομένα, να ε, έχουμε μια τέτοια επιχειρηματική νοοτροπία. Καλύτερο θα ήταν όμως να το έχουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι αλλιώς ο κατακαιρματισμός θα δυσκολέψει πολύ τα πράγματα. πώς ε, θα πετύχουμε τη συμμετοχή όλων των ε, ενδιαφερομένων. Ε, δύσκολο είναι, αλλά έχει γίνει τεράστια αλλαγή τα τελευταία πέντε χρόνια. Έρχονται επιχειρηματίες σε μένα και λένε ότι πρέπει να νομοθετήσετε. Ε, Προφανώ κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι αναπόφευκτο, άλλοι όμω λένε επίση ότι καλύτερα να κάνουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή, διότι νιώθουν και εκείνοι ότι οι πολίτε θα χάσουν την εμπιστοσύνη του στην τεχνολογία. Και βλέπω πώς οι επιχειρήσεις ε, αναλαμβάνουν πιλωτικό ρόλο. Από αυτά που μας έδωσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων λάβαμε 350 απαντήσεις πολύ, πολύ ψηλής ποιότητας ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών ε, των ηθικών αρχών. Είναι σημαντικό λοιπόν να ακούσουμε τις αντιδράσεις ε, και πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να γίνει ε, σωστά αυτό και δεν επιτρέπεται να υπάρξει αντίθεση ανάμεσα στους νομοθέτες και τις επιχειρήσεις και να ε, είναι στριμωγμένοι ανάμεσα τους οι πολίτες. Τέλος, όσον αφορά το θέμα μιας ανοιχτής σειράς κανόνων και το θέμα της δεοντολογίας, της ηθικής. Εμένα ε, με εμπνέει πολύ η δουλειά που γίνεται όσον αφορά την ε, επεξηγηματικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να εξηγεί η ίδια τι κάνει ε, ή να εξηγεί τι κάνουν ε, άλλα στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης, διότι και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί ένας αλγόριθμος ε, και ιδιαίτερα όταν έχουμε τεχνολογία που μαθαίνει, δηλαδή ξεκινάμε από ένα σημείο εκκίνησης, ε, γίνονται διάφορα πράγματα ε, και έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, υπάρχει ο κίνδυνος των μαύρων κουτιών, να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό το explainability. Είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε ε, να μην είναι απαραίτητο ο ίδιος ε, ε, επιστήμονας να είναι στην ίδια επιχείρηση όλα του τα χρόνια, διότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Υπάρχουν λοιπόν πολλά επίπεδα ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εάν όμως θέλουμε να εξετάσουμε θέματα ασφάλειας, ευθύνης, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να ασκήσει κανείς τα δικαιώματά του, διότι είναι πιο δύσκολο να καταλάβει κανείς τι πήγε στραβά όταν έχουμε τεχνολογίες που μαθαίνουν. Γι' αυτό θα πρέπει να επανεξετάσουμε την ε, ισχύουσα νομοθεσία για να διαπιστώσουμε αν πράγματι ε, είναι εφαρμόσιμη. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος είπε ότι πρέπει να έρθουμε και όταν ο πρόεδρος λέει κάτι πρέπει να το κάνεις. Μία ερώτηση μόνο ο καθένας από τους πέντε. Διότι εδώ είχαμε 20 πάνω κάτω. Ισμαήλ Αντούκ, Μαρία Μαρκές. Very short and Πολύ σύντομα. Και οι υπόλοιποι θα μιλήσω με τον ΣΕΠ και τον ΩΣΑ που είναι μαζί μας. Και θα έχουμε και άλλη τέτοια εκδήλωση. Ισμαήλ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το χρόνο. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε που ήρθατε και που μένετε λίγο περισσότερο. Ο πρόεδρος της Google είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πιο σημαντικό από την ηλεκτρική ενέργεια και τη φωτιά και θα δημιουργήσει ευκαιρίες τεχνητή νοημοσύνη, αλλά υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι, προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού. Ένα από αυτά είναι η αύξηση ανισοτήτων και έμφυλη ε, ανισότητα, δηλαδή μεταξύ ανδρών γυναικών και ανισότητες στην αγορά ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αρχή, εποπτικός φορέας που θα εξασφαλίζει την εποπτεία, ε, θα αποφύγει αυτά τα προβλήματα, θα είναι αποτελεσματικό εργαλείο ή θα συνεχίσετε να αφήνετε τις ιδιωτικές πλατφόρμες να αυτορυθμίζονται. Ποιες οι απόψεις σας όσον αφορά τα δεδομένα σαν δημόσιο αγαθό και πώς θα μπορεί να υπάρχει επιμερισμός αυτών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Μαρή Μαρκές, ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομη θα είμαι, χωρίς πολλές ευχαριστήσεις. Τι σκέφτεστε για πολιτική ανοιχτή όσον αφορά τα δεδομένα που έχουμε ενθαρρύνει σε διάφορες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα. Αν είναι πολύτιμη πηγή, πλούτος τα δεδομένα, μήπως πρέπει να εξεταστεί η πολιτική για τα ανοιχτά δεδομένα, τα ελεύθερα δεδομένα. Και όσον αφορά τον κοινό χώρο δεδομένων στον τομέα της υγείας περιπίνης, τι σκέφτεσαι στην Ευρώπη. Λοιπόν, μεγαλύτερη παραγωγή δεδομένων και επιμερισμό δεδομένων. Αλλά πρότυπα και προδιαγραφέ για τα δεδομένα. Αυτά που ε, έχουμε τώρα δεν μπορούν να μπουν σε αλγόριθμου, δεν είναι κατάλληλα. Μήπω θα πρέπει να έχουμε προδιαγραφέ και, στοιχεία, ε, και διάφορα επίπεδα στα οποία θα πρέπει να είναι τα δεδομένα. Είπατε ότι για να φτάσουμε να επιτύχουμε αυτήν την αριστεία χρειαζόμαστε και πόρους, χρηματοδότηση, χρειαζόμαστε όμως ε, και δεδομένα. Ξέρουμε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια και μεγάλες επενδύσεις στην Κίνα και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουμε και εμείς την Digital Europe. Πιστεύετε ότι αυτά που γίνονται στην Ευρώπη είναι αρκετά έτσι ώστε να βρεθούν οι καλύτεροι, οι άριστοι, ε, αυτοί οι οποίοι θα μας οδηγήσουν ε, στην κατάσταση που θέλουμε. Δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα στην έρευνα. Συνάδελφος εκεί πίσω παρακαλώ. Ας ακούσουμε λοιπόν τις απαντήσεις σας και υποσχεθήκατε, το λαμβάνουμε υπόψη, υποσχεθήκατε ότι θα επανέλθετε. Δεσμευτήκατε. Δίκιο έχετε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ε, μεροληψίας διότι μπορεί τα δεδομένα, οι ομάδες δεδομένων να έχουν κάποια απόκληση και για κάποια πράγματα δεν έχουμε δεδομένα. Και για μερικά πράγματα δεν έχουμε επαρκείς γνώσεις. Σε πολλές χώρες δεν έχουμε καν στατιστικά στοιχεία για τις αμοιβέ, για τα ημερομίστια, ανάλογα με το φύλλο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρέπει να βελτιώσουμε πολύ την ποιότητα των δεδομένων. Και θα πρέπει να επιβάλλουμε το επιθυμητό και το ευκταίο. Πώς, δεν ξέρω ποια θα είναι η δομή γι' αυτό. Είναι σημαντικό να μπορούμε να επιβάλλουμε αυτά που πρέπει να επιβάλλουμε για να έχουμε ε, τα δεδομένα που θέλουμε. Πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες καταρχάς, να τις εφαρμόσουμε. Καλύτερα απλές προτεραιότητες ξεκάθαρες παρά να έχουμε πολλές που δεν μπορούμε να επιβάλλουμε. Τώρα, τα δεδομένα στο δημόσιο αγαθό. Είμαστε εδώ 5-10 χρόνια. Από την αρχή ήταν καλό που είχαμε την πολιτική να διαθέτουμε τα δεδομένα σε μεγάλες ποσότητες για να καινοτομούν οι επιχειρήσεις. Δεδομένα για ποτάμια, ριάκια, υψόμετρα κλπ. Δορυφορικά στοιχεία. Αυτό που δημιουργούμε τώρα είναι το αντίστοιχο νέα γη. Σαν να έχουμε ανακαλύψει νέα γη. Σαν να έχουμε ανακαλύψει ορυχείο με νέο πλούτο ένα νέο μέταλλο που δεν είχαμε πριν. Αν φανταστείτε με τέτοια ανακάλυψη, τι κάνετε τότε. Λέτε όποιος έχετε πρώτος τον κύριο Νίδε. Δεν νομίζω. Θα έπρεπε να εξασφαλίσετε αυτός ο πόρος να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για καινοτομία, για επιχειρηματίες, για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες βέβαια. Κυρίως αν ο πολίτης είναι ο φορολογούμενος που πλήρωσε για να δημιουργηθεί αυτός ο πόρος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρετηθούμε από την ανοιχτή προσέγγιση στα δεδομένα, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία που παράγονται με χρήματα φορολογουμένου δίδουν και κάποια ωφέλη στο φορολογούμενο. Ας σκεφτούμε άλλους πόρους. Δεν θα αντιμετωπίζαμε άλλους πόρους όπως τα δεδομένα. Και υπάρχει μια έννοια στην αγορά. Αν έχεις πρόσβαση στα αγαθά, στα, δεδομένα και παράγει μια υπηρεσία και είσαι επιτυχή, τελικά θα κατακτήσει την αγορά για μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Λοιπόν, αυτό που έρχεται δεύτερο μετά από σένα, ίσω να είναι επιτυχή για να παράξει την, την υπηρεσία, αλλά δεν θα είναι επιτυχή στην αγορά, διότι ήδη έχουν μπει στο οικοσύστημα του πρώτου. Και αυτό δεν αρκεί να πούμε ότι ο καθένα μπορεί να ξαναχρησιμοποιεί τα δεδομένα και να κάνει το ίδιο όπω ο πρώτο, διότι υπάρχουν και συνέπειε αγορά το πώς χρησιμοποιούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κουβεντιάσουμε αυτό τώρα, διότι θα αλλάξει ο ρυθμός όσον αφορά την παραγωγή δεδομένων λόγω του διαδικτύου των πραγμάτων, Internet uh, of Things, και οι κυβερνήσει θα είναι πιο ψηφιοποιημένε και θα παρέχουν περισσότερε υπηρεσίε ψηφιακά. Και γι' αυτό περισσότερα δεδομένα με τη σειρά του θα παράγονται. Έξοχο αυτό. Αυτό που υπόθηκε, ότι χρειαζόμαστε πρότυπα και προδιαγραφέ κυρίως αν θέλουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να συμμετέχουν. Πιθανότατα θα ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ειδική πρόσβαση σε δορυφορικά στοιχεία. Κυρίως φροντίζουν αυτά τα δεδομένα της μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα. Και αυτό διότι έχουν πρότυπα, συμμορφώνονται με πρότυπα και ξέρουν πώς να προσεγγίσουν το όλο θέμα. Βέβαια, ε, μπορεί τώρα να έχει την τεχνολογία που να βρει και βελόνα στα χείρα, και χρειάζεται η τεχνολογία για να βρει βελόνα στα χείρα. Εάν θέλεις ε, πιο μεγάλη πρόσβαση, πρέπει να διοργανώνει τα στοιχεία με ένα τέτοιο τρόπο που να είναι πιο προσβάσιμα. Νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε κοινού χώρου δεδομένων. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ επικοδομητικό και μπορεί να δημιουργήσει εμπιστοσύνη για τη χρηματοδότηση. Η Ευρώπη είναι έξοχη όσον αφορά την παραγωγή γνώσης και τεχνητής νοημοσύνης. 30% των ακαδημαϊκών μελετών για τεχνητή νοημοσύνη προέρχονται από την Ευρώπη. Στην τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσεται μεταξύ επιχειρήσεων έχουν πολλά να προσφέρουμε, αλλά έχουμε πολύ λίγα χρήματα. Δεν αφορά μόνο εμά σαν Ευρώπη, αλλά και τα κράτη-μέλη αφορά το θέμα. Τα κράτη-μέλη δεν επενδύουν αρκετά στην τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς βέβαια ελπίζουμε ότι με τον ορίζοντα Ευρώπη, Horizon Europe και με την ψηφιακή Ευρώπη και τα διάφορα προγράμματα Digital Europe μπορούμε αυτό να το βελτιώσουμε και να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις και έτσι ελπίζουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες για διαπραγματεύσεις για τον επόμενο επταετή προπολογισμό για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα διαπιστώσουμε και θα καταλάβουμε να επενδύσουμε στο μέλλον. Δεν θέλω αυτό να... να πω ότι είναι ένας αγώνας, αλλά είναι αγώνας και πρέπει να προσελκύσουμε ταλέντο και να χρησιμοποιήσουμε στο βέλτιστο βαθμό την ε, τεχνογνωσία. Όχι λόγω γεωπολιτικών παραγόντων, διότι διαφορετικά δεν θα υπηρετήσουμε όπως πρέπει τους ε, πολίτες. So, I think the future... Νομίζω ότι το μέλλον βρίσκεται σε καλά χέρια, διότι έχετε γνώσεις, έχετε όραμα, και όσον αφορά τον αγώνα αυτόν θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Θα συνεχίσουμε εμείς τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Εμείς θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. I'll take the rest of the questions that... Θα ακούσουμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις. προς τους ομιλητές μας. Έχουμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για να διαμορφώσουμε τις πολιτικές μας. Ε, τον Άντωνη Γκούτς, ε, που είναι Διευθυντής ε, Δημοσίων Σχέσεων στον ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ δημιουργεί και εφαρμόζει παγκόσμια πρότυπα. Είδαμε λοιπόν ότι ο Άντωνη το έχει καταφέρει αυτό επανειλημμένα με τα ε, εργαλεία για τον ε, ψηφιακό φόρο, με ε, το blockchain, την τεχνολογία λυσίδασης στοιχειών και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουμε μαζί μας και τον και πολύ σημαντικό σύμβουλο για τις εργασίες του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ρέντα. Ε, δεν ξέρω αν θέλουν να κάνουν κάποια εισήγηση πρώτα ή ε, θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις πρώτα. Παρακαλώ. Άντωνη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Εύα, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το Δεκέμβριο του 2018 ήμουνα τελευταία φορά εδώ για μια εκδήλωση και βλέπω το ότι Παρά την 45 λεπτή καθυστέρηση είναι πολύ ε, δημοφιλής αυτή η εκδήλωση. Ε, καταλαβαίνετε πόσο συγκινημένος νιώθω, διότι από την προφορά μου καταλαβαίνετε ότι είμαι μισός Βρετανός και μισός Ισπανός. Εργάζομαι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και 14 χρόνια και και έχω ασχοληθεί και με ε, την ε, την διαδικασία αυτή. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Πάντως ε, σημαντικό είναι ότι ακόμα κι αν ήμουν μόνο Βρετανός, αποκλειστικά Βρετανός, στον ΩΣΑ θα μπορούσα να συνεχίσω να συνομιλώ μαζί σας. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι καθαρά εγωιστική. Καταλαβαίνω ότι έχουμε εδώ ε, ανθρώπους ε, με μεγάλη επιρροή η εγωιστική μου λοιπόν ε, παρατήρηση ε, απευθύνεται και σε εσά. Ο ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Και νομίζω ότι ε, θα γνωρίζετε κάποια από τα πράγματα που έχουμε κάνει και θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά. Θα ήθελα να σας ζητήσω να Συνεργαστείτε μαζί μα διότι βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Ε, πρέπει λοιπόν να αφουγκραστούμε. Αυτό είναι το ε, κομμάτι τη επικοινωνία ε, που προκαλεί τι περισσότερε δυσκολίε στου ανθρώπου. Να μην υποθέσουμε λοιπόν ότι γνωρίζουμε τα πάντα, ότι γνωρίζουμε ποιε είναι οι βασικές ανησυχίες και ελπίδες των ανθρώπων. Πώς μπορούμε να το μάθουμε αυτό. Εγώ από το 2008 συμμετέχω στον ε, ΟΣΑ, είχαμε την ε, παγκόσμια οικονομική κρίση και παρόλα αυτά δεν είχαμε επαφές με τους νομοθέτες. Η δουλειά μας ε, είναι καλύτερες πολιτικές και καλύτερες ζωές. Αυτό δεν είναι απλά ένα σύνθημα. Ποιος τα κάνει αυτά καλύτερα, εσείς. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε επαφή με νομοθέτες και βουλευτές περισσότερο από ποτέ και θεωρώ ότι οι επαφέ μεταξύ μα θα είναι πολύτιμε και για εσά. Και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στην περίπτωση τη τεχνητή νοημοσύνης. Είναι μια τεχνολογία γενικού σκοπού. Τι σημαίνει αυτό, ότι επηρεάζει τα πάντα. Είναι σαν την τεχνολογία λυσίδα συστοιχειών, το blockchain. Η Εύα και εγώ γνωριστήκαμε όταν ε, μιλούσαμε για το, για το blockchain. Ε, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχει να κάνει μόνο με ε, κρυπτονομίσματα, αλλά όχι και τώρα, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, πολλοί ίσω νομίζουν ότι αφορά μόνο τα, την αυτόνομη οδήγηση, τα αυτοκίνητα χωρί οδηγό. Σε πολλούς τομείς λοιπόν βλέπουμε να εμφανίζονται ε, τεχνολογίες. Πραγματικά δεν θα ήθελα να βρίσκομαι στη θέση της Επιτρόπου Βεστάγκερ. Ε, την εμπιστεύεστε. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δημιουργούμε εμείς την πρώτη ομάδα για την τεχνητή νοημοσύνη με παγκόσμια εκπροσώπηση βουλευτών στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού δικτύου του ΟΣΑ και θα συναντηθούμε πρώτη φορά στις 26 Φεβρουαρίου ε, στο Παρίσι. Η Εύα το γνωρίζει, αυτό είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη, συμμετέχει στο δίκτυο εδώ και πολλά χρόνια, την ενδιαφέρουν πολύ τα φορολογικά θέματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και είναι ιδιαίτερα επίκαιρα αυτή τη στιγμή. Όλοι θα έχετε ακούσει για τον ψηφιακό φόρο και συνδέονται αυτά μεταξύ τους. Ιδιαίτερα το θέμα των πόρων που έθιξαν πολλοί από εσά. Ε, τι πόρους έχουμε στη διάθεσή μα, έχουμε επαρκείς πόρους. Ε, το να πετύχουμε συμφωνία πάνω στη φορολογία συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ε, θα είναι ένας ε, ενάρετος κύκλος, διότι θα μπορέσουμε έτσι να ελέγξουμε τα θετικά στοιχεία, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε προστασία αφενός και να τα αναπτύξουμε περαιτέρω. Καλό λοιπόν ε, το, τους ευρωβουλευτές, ε, το προσωπικό του Κοινοβουλίου και άλλους ενδιαφερομένους ε, να συμμετάσχουν μαζί μας στην προσπάθεια αυτή. Είμαι βέβαιος ότι θα οργανώσουμε και συναντήσεις της ομάδας αυτής εδώ στο Κοινοβούλιο στο μέλλον. Σε ευχαριστώ, Άντωνη. Αντωνή Κόχ είναι εδώ και βεβαίως έχουμε και τον άλλο καλεσμένο μας. Θα ήθελα να ακούσω και την δικιά σας άποψη και τώρα και στο μέλλον. Οπωσδήποτε θα έχουμε επαφή και στο μέλλον, αλλά πρώτα να σας, ακούσω, να σας ακούσω και μετά θα πάρουμε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούει κανείς την Αντιπρόεδρο Φερστάκερ. Το όραμα που έχει ε, αποτελεί πηγή έμπνευσης ε, για όλους αλλά και μεγάλο στοίχημα. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι υπάρχει όμως και ένα θέμα ουσίας πίσω από όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ε, συγκρίσεις σχετικά με το πόσο επενδύουμε σε αυτό το τομέα ή πόσο σε άλλους. Η τεχνητή νοημοσύνη από την φύση της είναι επεκτατική, πράγμα που σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε απόφαση ε, πάρετε στο μέλλον ε, για έρευνα, για νομοθεσία, για ε, οτιδήποτε άλλο, η τεχνητή νοημοσύνη οπωσδήποτε θα εμπλέκεται. Επίσης, η Επίτροπος, στα πλαίσια της νέας Επιτροπής, εργάζονται με μια δέσμευση την οποία αποκαλούν γεωπολιτική δέσμευση. Άλλωστε, έχουν προχωρήσει και στην λεγόμενη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Green Deal. Ε, κοιτάξτε, μιλάμε για κάτι το οποίο προέρχεται από την Επιτροπή και το οποίο ε, για την επόμενη δεκαετία θα έχει μια χρηματοδότηση, μια μόχλευση οικονομική που θα φτάνει τα 400 δις κλπ. Πάντως έχουμε ε, μεταβάσεις. Η μία είναι η οικολογική και η άλλη είναι η ψηφιακή. Οι δύο αυτές μεταβάσεις θα πρέπει να ειδωθούν από κοινού. Ε, γιατί ξέρετε οποιαδήποτε μετάβαση ας πούμε σε σχολικό περιβάλλον μπορεί να είναι επικίνδυνη αλλά ξέρετε και κάθε είδος τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι εξίσου σημαντικό. Κάθε είδους τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απαραίτητο να προωθηθεί κατά την δική μου άποψη και αυτό το κατάλαβα πολύ νωρίς ε, όταν ασχολήθηκα με το υψηλού επίπεδου ε, τμήμα, την υψηλού επίπεδου ομάδα της Κομισιόν ε, για την τεχνική, τεχνητή νοημοσύνη, κατάλαβα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τα θέματα από δεοντολογική άποψη, αλλά και από την άποψη και την οπτική γωνία της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει την τεχνική νοημοσύνη ως σκοπό ή αυτοσκοπό. Πρέπει να τη χρησιμοποιήσει ως μέσον. Ε, δεν είναι μόνο για να βγάζουμε selfies και να λέμε τι ωραίοι που είμαστε ή να βάζουμε φιλτράκια για να γινόμαστε πιο όμορφοι. Ε, πρέπει να μπορέσουμε να επενδύσουμε ας πούμε πόρους για την τεχνική νοημοσύνη για άλλα πράγματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε ή να προσεγγίσουμε τους ε, ε, στόχους βιωσιμότητας. Ε, θέλουμε, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πόροι για την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έχουμε αυτό το το ε, κτίνος απέναντί μας, το οποίο με κάποιο τρόπο το θηρίο πρέπει να το δαμάσουμε. Πρέπει να βρούμε τρόπους ε, να δαμάσουμε λοιπόν το θηρίο αυτό. Εγώ δεν θέλω να φανώ παλιωμοδίτης ή να ακουστώ παλιωμοδίτης, ε, αλλά εάν δείτε το μοντέλο ας πούμε που μας δίνει η κινέζικη κοινωνία με μια τεχνητή νοημοσύνη χωρίς όρια, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, τότε πραγματικά βλέπουμε ότι είναι ένα κακό μοντέλο Έχουμε δει κάποια προφανή στην ε, ε, Κίνα. Από την άλλη μεριά βλέπουμε και στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, αύξηση των ανισοτήτων. Βλέπουμε να ανθούν εντός εισαγωγικών οι ανισότητες στη χώρα της Silicon Valley. Και μάλιστα το είπε προηγουμένως η Αντιπρόεδρος ότι δεν είναι όλες οι καινοτομίες, οι καινοτομίες ισότητας. Πρέπει λοιπόν να τα ξεχωρίσουμε αυτά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι τεχνητή νοημοσύνη θέλουμε, γιατί πολλές φορές λέμε χάσαμε το τρένο της καινοτομία, χάσαμε το τρένο της ανάπτυξης, δεν θα τα καταφέρουμε. Όχι, αλλά πρέπει να τα ξαναδούμε λίγο αυτά. Νομίζω ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσείς, οι εμπειρογνώμονες, οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν το απαραίτητο, ε, τον απαραίτητο κοινό τόπο, τη χρυσή τομή, έτσι ώστε ε, να διασφαλιστούν όλοι οι ε, στόχοι. Εγώ είμαι ακαδημαϊκός και ε, η ακαδημαϊκή ύλη μας λέει ότι η συμπληρωματικότητα της καλής νομοθεσίας, της καλής ρύθμισης με την σωστή καινοτομία μπορεί να δώσει αυτό το απαραίτητο, τον σωστό απαραίτητο μέσο όρο. Δεν πρέπει να ε, δημιουργήσουμε μια τεχνητή νοημοσύνη ή μάλλον να το πω διαφορετικά θα πρέπει να σχεδιάσουμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το κάνει γιατί κατανοεί ε, καλύτερα από άλλες περιοχές του κόσμου τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, εμείς νομίζω ότι καταλαβαίνουμε καλύτερα από άλλους ότι μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο όμως δεν θα σταματήσει σταματήσει την καλή τεχνητή νοημοσύνη. Θα σταματήσει μόνο την τεχνητή νοημοσύνη που δεν θέλουμε και θα οδηγήσει εν τέλει την τεχνητή νοημοσύνη στις κατευθύνσεις που εμείς επιθυμούμε. Ως ακαδημαϊκός λοιπόν και ως think tanker, ως συμμετέχον σε ομάδες προβληματισμού, αυτά έχω να σας πω. Κοιτάξτε, κανείς δεν κατέχει την τέλεια συνταγή. Όλοι έχουμε ευθύνες, δεν όχι τόσο μεγάλες όσο εσείς που είστε στο κοινοβούλιο ή εσείς ε, η Αντιπρόεδρος στην Κομισιόν ή ακόμα και ο Άντωνη. Εγώ όμως ε, θα είμαι πάντα στο πλευρό σας και θα συμβάλλω έτσι ώστε ε, να κατανοήσουν όλοι ότι το τρένο των δεδομένων όχι μόνο δεν το έχουμε χάσει, αλλά δεν έχει καν φύγει ακόμα από το σταθμό. Με, αυτό το πνεύμα θα πρέπει να μιλήσουμε στον υπόλοιπο κόσμο, θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και τις μηχανές και ανάμεσα στον πλανήτη και τις μηχανές. Uh, λοιπόν, όλο και περισσότεροι επιφανείς βουλευτές έρχονται και συμμετέχουν στη συζήτηση. Είναι η αρχή τώρα και για μας για το Κέντρο Τεχνητός, Τεχνητής Νοημοσύνης και της στοά για πρώτη φορά να μπορούν να συντονίζονται και να θέσουν καλά πρότυπα για την ψηφιακή εποχή είναι πολύ σημαντικό. Όσα βοηθάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ηνωμένα Έθνη είναι η μεγάλη επέκταση, η μεγάλη φορή θα προσπαθούμε να έχουμε εδώ, γιατί το 2020 είναι η χρονιά που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε γενικές προδιαγραφές, ούτως ώστε αυτή ε, η τεχνολογία να πλησιωθεί σωστά. Ο κύριος Έλερ, η αντιπρόεδρος κυρία Μαγκίνες, είναι μαζί μας. Μεγάλη τιμή, όπως σας είπα, είναι ιστορική ημέρα, δεν είναι εύκολη ημέρα αλλά ίσως είναι σημαντικό να ξεκινήσει η συζήτηση για το μέλλον σήμερα. Όποιος επιθυμεί να μιλήσει από τους συναδέλφους πρώτος, ορίστε. Εσύ, ευχαριστώ για ε, την όλη παρουσίαση και που είσαστε εδώ. Θα ξέρετε ίσως ότι υπάρχει ένα σχέδιο λευκής βίβλου. Κάπου υπάρχει, κάπου βρίσκεται. Όμως, κατά την άποψή μου είναι αρκετά καλό έγγραφο. Περιγράφει το τοπίο. Δεν προτείνει συγκεκριμένα πράγματα και νομοθετικές αποφάσεις, όμως αναφέρει επιλογές. Τρεις βασικά είναι οι επιλογές. Πρώτα, εθελοντική ετικεταθεσία. Δεύτερη, τομιακές απαιτήσει τονίζονται στην αναγνώριση προσώπων. Το τρίτο, να εντοπιστούν οι τομεί υψηλού κινδύνου και να αντιμετωπιστούν πρωτίστω. Από ό,τι ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζεται περισσότερο ή προτιμάει την τρίτη επιλογή. Αν εσείς έπρεπε να αποφασίσετε, τι προσέγγιση θα ακολουθούσατε έναντι των τριών αυτών επιλογών. Ευχαριστώ. Δεύτερος, θα ακούσουμε τους αντιπροέδρους της ΣΤΟΑ. Κρίστιαν. Ίσως επειδή είμαι Γερμανός, ακολουθώ πρακτική προσέγγιση. Διαπραγματευόμαστε στο, τον προπολογισμό στο τέλος του έτους. Έχουμε δύο πόρους για χρηματοδότηση, για δημόσια χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα έχουμε το πρόγραμμα πλαίσιο. 15 δις ευρώ έχουμε για ψηφιακή τεχνολογία και διάστημα εν γέννη. Και μετά έχουμε 16 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα για Connect, για τη Ευρώπης. Εκεί έχουμε περίπου 2,5 για τεχνητή νοημοσύνη. Τα υπόλοιπα θα βγουν από το πρόγραμμα πλαίσιο. Ίσως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων υπάρχουν κάποια χρήματα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα δημοσία λέμε ότι θέλουμε να ξοδέψουμε 1,5 δις το χρόνο για τεχνητή νοημοσύνη. Με απλούς υπολογισμούς δεν χάσαμε στη τεχνητή νομοθεσίνη. Αν έχετε 2,5 στο Connect, τα 8 δις θα πρέπει να βγουν από το ψηφιακό. Αν δείτε τις αναλογίες μεταξύ διαστήματος και ψηφιακού τομέα, στο, πλαίσιο, στο πρόγραμμα πλαίσιο περίπου 4 δις με 5 δις θα πάνε στο διάστημα. Αυτή είναι η ποσόστοση ιστορικά και 10 δις μένουν. Πρακτικά 90% αυτού θα πάει στην τεχνητή νοημοσύνη. Εξού και ερώτησή μου. Τις αναλογίες πώς τις βλέπετε. Θέλουμε να κινηθούμε και στον τομέα της κβαντομηχανικής τους υπεροϋπολογιστές αν κατασκευάσουμε μέσω κβαντικής τεχνολογίας και έχουμε διάφορα θέματα. Πώς θα μοιράσουμε τις φιλοδοξίες. Ανησυχώ κάπως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ανακοινώνει 10,5 δις ή 11 και στην πράξη δεν ξέρουμε το Συμβούλιο θα μας δώσει αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και αντιρρήσει του προπολογισμού. Έχουμε τη σημασία τη τεχνητής νοημοσύνη από τη μια και τι άλλε φιλοδοξίε, κβαντική τεχνολογία κλπ. Συναφή θέματα όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Και άλλη ερώτηση. Η κυρία Βεστάγκερ αναφέρθηκε στη σημασία των δεδομένων. Τα δεδομένα παράγονται με δημόσιο χρήμα. Αυτά πρέπει να θεωρηθούν κάτι, σαν κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό. Τα δεδομένα τα βλέπουμε στα πλαίσια τεχνητής νοημοσύνης και λογαρίθμων. Αλλά εντάσσονται και σε άλλα συστήματα. Είπε η κυρία Βεστάγκερ ότι πρέπει να προσέχουμε για την χρήση των δεδομένων. Είχαμε πάντα πολιτική ανοιχτών δεδομένων και τώρα μάλλον θα πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση και προβλέπουμε ότι Θα πρέπει η κοινωνία χρησιμοποιεί τα δεδομένα, να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την ευρύτερη κοινωνία. Αυτό ήταν πριν. Ξέρουμε όμως οι μεγάλες εταιρείες ρουφάνε τα δεδομένα που παράγουμε εμείς δωρεάν και τα απορροφάει η Google και τα χρησιμοποιεί και άλλοι. Το open, open, open, ανοιχτά, ανοιχτά, ανοιχτά, αυτή η ιδεολογία είχαμε πριν. Από την άλλη, λέει η κυρία Βεστάγκερ, πληρώσαμε για την παραγωγή δεδομένων, αλλά πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά ποιο θα ωφεληθεί, ποιο θα πάρει τα δεδομένα. Τα δεδομένα ε, που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα για την έρευνα με 120 δις Φερρυπίν. Η Αντιπρόεδρος Μακίνας. Έχετε ερώτηση? thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ζήτω συγγνώμη που καθυστέρησα. Ήταν δύσκολη μέρα σήμερα. Η ερώτησή μου δεν θα είναι ευφυής, διότι δεν γνωρίζω το θέμα αυτό. Ε, έχει να κάνει όμως με τη ρύθμιση. Μερικές φορές εδώ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ρυθμίζουμε, όταν νομοθετούμε, είμαστε καχύποπτοι όταν έρχονται άνθρωποι από τον οικονομικό τομέα. Ε, εγώ όχι. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές οι επαφές. Ε, ε, μπορείτε να μας καθοδηγήσετε, διότι χρειαζόμαστε ανθρώπους που να ασχολούνται με τα θέματα αυτά, που να έχουν τις γνώσεις, ε, τις δεξιότητες ε, και χρειαζόμαστε τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να νομοθετήσουμε. Μπορούμε να έχουμε τέτοιες επαφές, μπορούμε να πληρώσουμε για να το έχουμε αυτό και... Ε, δεν είναι πολύ εύκολη η επαφή αυτή. Ευχαριστώ, κυρία Νάτα. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου είναι νομίζω μια ανησυχία πολλών. Ως γυναίκα, Ως γυναίκα πολίτης, ε, πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για τα θέματα ηθικής. Ε, άκουσα ότι ασχολείστε με αυτά και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ε, ηθικές κατευθυντήρες γραμμές. Η δική μου ανησυχία είναι ότι γνωρίζουμε ότι σε διάφορες χώρες υπάρχουν διαφορετικά ηθικά δεντολογικά πρότυπα. Όταν είμαστε όλοι υπερσυνδεδεμένοι δεν θα μπορέσουμε να ε, θέσουμε σύνορα στην εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, σε όλες τις διαδικασίες όπου θα λαμβάνονται αποφάσεις. Πώς μπορούμε να βρούμε τρόπο να ελέγξουμε τις επιπτώσεις ε, αποφάσεων που λαμβάνονται με βάση άλλα ηθικά πρότυπα. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι... Ακούσα ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη ε, να οδηγήσει σε ε, συσκευές με συνείδηση. Μια τέτοια συσκευή, αν κάποια μέρα θεωρήσει ότι οι άνθρωποι είναι άχρηστοι, και ότι αποτελούν πρόβλημα για την ανάπτυξη του κόσμου, τι θα γίνει τότε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και θα ήθελα να προσθέσω ότι καθότι έχουμε τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, ε, είχαμε εδώ μια πολύ ισχυρή πρωτοβουλία την προστασία του ιδιωτικού βίου. Άκουσα την ε, κυρία Βεστάγκερ που έλεγε ότι δεν, θέλουμε, δεν θέλει να αλλάξουμε τον ε, κανονισμό. Θέλουμε όμως να τον ενισχύσουμε διότι το opt-out δεν ε, οδηγεί σε ευαισθητοποίηση. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε opt-in, να επιλέξουμε να συμμετάσχουμε ε, και να προστατεύσουμε τα ευαίσθητά μας δεδομένα. Ε, θα ήθελα το μικρόφωνο, ε, το τηλέφωνο μου, η φωτογραφική μου μηχανή να κλείνουν όταν δεν τα χρησιμοποιώ, διότι δεν έχω τη δυνατότητα αυτή. Μήπως θα πρέπει να υπάρχει η υποχρέωση ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι ε, δεδομένα συλλέγονται και όλοι έχουν στα χέρια τους τη λευκή βίβλο Ναι, εντάξει, είναι μυστικό, αλλά όλοι το γνωρίζουν. Ε, αναφέρεται στο ανατομέα. Πιστεύετε όμως ότι ανατομέα ή αναχρήση θα πρέπει να γίνονται αυτά. Θα δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον Άντωνη και κατόπιν στον Ανδρέα. Εγώ θα το έλεγα ανάποδα. Ίσως δεν έχω, δεν έχω διαβάσει τη Λευκή Βίβλο, ίσως είμαι και ο μόνος αλλά υπάρχουν ε, κάποια ερωτήματα επί των οποίων θα ήθελα ε, να απαντήσω μετά από τον Ανδρέα. Ναι, ναι, έχω διαβάσει εγώ τη Λευκή Βίβλο και το ομολογώ ένοχος ο κατηγορούμενος. η Κομισιόν ε, στο τέλος του, της Λευκής Βίβλο λέει ποιες θεωρεί πιο βιώσιμες λύσεις και εναλλακτικέ. Πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για ανοιχτή διαδικασία. Τώρα θα γίνει και μία αξιολόγηση αντικτύπου, ε, θα γίνει ανάλυση όλων των εναλλακτικών. Αυτή είναι η διαδικασία που ήθιστε να ακολουθούμε από την στιγμή που θέλουμε κάποια βίβλος, λευκή βίβλος, να ε, γίνει εν τέλει νομοθεσία. Και βεβαίως ε, θα ξεκινήσει και ακαδημαϊκή και επιστημονική συζήτηση. Τώρα, η ιδέα ενός συστήματος πιστοποίησης, certification system, φαίνεται μάλλον περίπλοκη προς ώρας τουλάχιστον. Θα δούμε ε, τι θα γίνει. Θα πρέπει ε, να έχουμε βασικά τις πρώτες δεοντολογικές ηθικές αρχές και τις αντίστοιχες ε, νομοθετικές διατάξεις. Ε, βεβαίως όλο αυτό το σύστημα χρειάζεται καλή διακυβέρνηση Υπάρχει και μία ιδιαιτερότητα σε αυτήν την ε, αγορά. Δεν είναι ότι, ε, είναι πολύ ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η ιδιαιτερότητα αφορά στην ε, ταχύτητα. δεν μπορούμε να βασιστούμε σε κάποια σώματα τα οποία θα μπορούν να ακολουθήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας. Θα πρέπει να είναι μάλλον κάποιο δίκτυο εθνικών ρυθμιστών ή εθνικών ρυθμιστικών αρχών με επίκεντρο ας πούμε την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή ο, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται το νομικό ε, πλαίσιο ε, θα είναι στην ουσία ένας χώρος στον οποίο δίνουμε σε αυτούς που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη πριν την εισάγουν στην αγορά να κάνουν αυτοαξιολόγηση με τρόπο όσο γίνεται πιο διαφανή ποιοι είναι τώρα οι ε, κίνδυνοι, αν θα είναι οι ίδιοι σήμερα και μετά από δύο εβδομάδες. Ε, κοιτάξτε, όταν ε, θα αναπτυχθούν αυτά τα προϊόντα στην αγορά, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν διαρκή επικαιροποίηση, έτσι ώστε να υπάρχει μετριασμός κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προκύψει ένας ενισχυμένος μηχανισμός διακυβέρνησης που μπορεί να έχει διάφορες μορφές, μπορεί να είναι κάποια δομή ε, πέρα και πάνω από την δομή προστασίας δεδομένων. Πάντως δεν είναι ένα σύστημα το οποίο ε, θα λειτουργεί μόνο του, θα δημιουργείται μόνο του. Αυτό είναι βέβαιο. Όσον αφορά τα open data, μάλλον όχι. Πρώτα η ερώτηση για τον προϋπολογισμό. Για μία ακόμα φορά λέω ότι δεν λέω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής ε, με το Fond Zero Mark για την ώρα. Το ζήτημα είναι ε, πώς ε, θα διαμορφωθούν ε, αυτοί οι προϋπολογισμοί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Εγώ αναμένω το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής πολιτικής, οι εταιρικέ σχέσεις, οι αποστολές να έχουν οπωσδήποτε ένα σημαντικό στοιχείο ή πεδίο τεχνητής νοημοσύνης. Σκεφτείτε όλες αυτές τις αποστολές που έχουν εντατική τεχνητή νοημοσύνη. Σκεφτείτε τις έξυπνες τις ε, πόλεις ε, ε, νομίζω ότι άλλωστε σε δύο χρόνια θα μιλάμε περισσότερο για το ίντερνετ των πραγμάτων παρά για την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, θα υπάρξει ε, ένα είδος ε, ήπια αιρεσιμότητα, soft conditionality όσον αφορά τα θέματα αυτά και όσον αφορά και τις τομεακές αρχές επί των οποίων θα σχεδιαστεί και θα λειτουργήσει η χρηματοδότηση. Το Horizon Europe θα συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε τους εμπειρογνώμονες και τους ε, επιστήμονες που θα είναι σε θέση να οδηγήσουν ε, στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί ήδη από την πρώτη σελίδα αναφέρονται οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης ε, και μετά να υπάρξει επαναπροσδιορισμός των στόχων. Αυτό είναι το μάντρα κατά κάποιο τρόπο της Κομισιόν. Είμαστε λοιπόν, ε, προσανατολιζόμαστε βάσει της ε, αποστολής και βάσει της ιδέας ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η βέλτιστη εκδοχή της τεχνολογίας. Επομένως, έρευνα, βασική έρευνα και εφαρμογή στην ε, ε βιομηχανία, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πόρων θα αφορά την τεχνική νοημοσύνη. Μετά τα open data, τα ανοιχτά δεδομένα, εγώ είμαι ελεύθερος στη σκέψη μου. Έχω μεγαλύτερες ελευθερίες από ό,τι περισσότεροι στην αίθουσα. Και έχω την αίσθηση ότι η ανοιχτή χρήση πάση θυσία ε, πέρασε. Μα τέλειωσε αυτό. Πάει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγε ανοιχτή καινοτομία, ανοιχτέ επιστήμε, ανοιχτή στον κόσμο. Πιο οικουμενική από τον Δαλάη Λάμα ή πνευματικό γκουρού. Το δοκιμάσαμε αυτό και ήταν άλλε εποχέ. Τώρα τα δεδομένα έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάποια δεδομένα, κυρίω αυτά παράγονται με δημόσιο χρήμα, πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για ερευνητέ, κυρίω. Δεν χρειάζεται να μεταμορφωθεί αυτό σε ένα μονοπόλιο δεδομένων. Η υποχρεωτική διαλειτουργικότητα αυτών των στοιχείων είναι μία από τι επιλογέ. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μεγιστοποιούν την αξία τους όταν παραμένουν ε, σε κοινή χρήση αλλά όχι ανοιχτά. Δεδομένα από το σύστημα ευρεσιτεχνιών έχει την μεγαλύτερη αξία όταν παραμένει εμπιστευτικό δεδομένο. Αυτό είναι διαφορετικό. Δεν λέμε όσο πιο ανοιχτά είναι τόσο καλύτερα. Το ανακαλύψαμε αυτό. Μας μαγνήτησε το διαδίκτυο επειδή δεκαετίες που είναι ανοιχτό πάση θυσία, τώρα πρέπει να πιστέψουμε στην πραγματικότητα. Και η βιομηχανική πολιτική εξωτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αφορά το μοίρασμα των δεδομένων, αλλά είναι σημαντικό και για άλλο λόγο το να μοιραζόμαστε δεδομένα και να παραμένουν στο βαθμό του δυνατού τα δεδομένα κλειστά, να είναι κοντά εκεί που παράγεται η αξία, η υπεραξία, είναι ένας τρόπος διαφύλαξης των βιομηχανιών μας και των χρηστών από τις ε, κεντρομόλες δυνάμεις που προσελκύουν τα στοιχεία στις πλατφόρμες. Και έχουμε έναν λόγο. Θέλουμε να εξισορροπήσουμε τα πράγματα. Θέμα βιωσιμότητας κοινωνική και οικονομικής διότι στην Ευρώπη αλλά και αλλού δεν μπορεί να προχωρήσει ισορροπημένα οικονομία αν αυτοί που παράγουν την υπεραξία δεν εισπράττουν κέρδη. Αυτό είναι σημαντικότατο. Θα μπορούσα να συνεχίσω αένα, αλλά δεν θα ήταν δίκαιο να έκανα κάτι τέτοιο. Το δεντολογικό στοιχείο και το GDPR για την προστασία των δεδομένων δηλαδή, η νομοθεσία, το GDPR έχει μια συνιστόσα που είναι και σχέδιο μελλοντικέ πρωτοβουλίε. Ε, Εξοδαφικό χαρακτήρα του GDPR. Και ίσω να κάναμε κάποια λάθη σε την νομοθεσία προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά μπορεί να διορθωθούν ίσω, να προσαρμοστεί το GDPR στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά με το GDPR έχουμε ένα κομμάτι σημαντικό που είναι υπόδειγμα τον υπόλοιπο κόσμο. Καλή αφετηρία για μα. Βοηθάει την ενιαία αγορά το GDPR. Και όποιο θέλει να έρθει σε επαφή με του Ευρωπαίου καταναλωτέ όπου και να βρίσκεται στον κόσμο. Πρέπει να συμμορφωθεί με το GPR αν θέλει να εισέλθει στην ενιαία αγορά. Και κάποια στοιχεία αυτού θα επηρεάσουν και την προσπάθεια να βάσουμε τον πύχη για υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι πρέπει να έχουν τα πράγματα. σω να δικαστικά να είναι πιο εύκολα τα πράγματα, πιο ευέλικτα, ίσω να είμαστε πιο ευέλικτοι και προσαρμοσμένοι. Το μελλοντικό σύστημα θα αντλήσει μαθήματα από την εποχή του GDPR και το GDPR 2, μορφή 2, θα είναι ακόμα εξοδαφικό, αλλά πιο ευέλικτο και θα μπορεί να προσαρμόζεται προθώντας τις αρχές που θέλουμε. Τέλος. Η αυτογνωσία, η αυτοσυνείδηση. Εγώ είμαι οικονομολόγος. Το πιο άχρηστο επάγγελμα στον κόσμο, κυρίως όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Επεξεργαζόμουν τεχνολογία επί σειρά ετών και πολιτική, αλλά βασίζομαι σε εμπειρογνώμονες. Όταν χρειάζεται να ξέρω κάποια πράγματα τόσο δύσκολα και ευαίσθητα, ρώτησα πολλού εμπειρογνώμων στην ερώτηση αυτή. Για την μοναδικότητα, την ε, αυτοσυνείδηση και το μήνυμα, πώς συνοψίζεται από αυτά που ρώτησα, η διαφορά μεταξύ εκείνων που μιλάνε για στενή τεχνητή νοημοσύνη και εκείνοι που μιλάνε για αποκλειστικότητα και μοναδικότητα είναι πολύ κοντά. Λένε είναι η διαφορά μεταξύ αστρονομίας και αστρολογίας μεταξύ των δύο. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο. Okay. Καλώς. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και μάλιστα έθιξε σε ένα θέμα που είναι δύσκολο να αναφερθεί. Στην Ευρώπη μιλάμε για ανοιχτή καινοτομία και τώρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει αμοιβαιότης. Η Κίνα προσπαθεί να εξασφαλίσει, να κλειδώσει στοιχεία και να τα κλειδώνει τοπικά στο διαδίκτυο. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την κυριαρχία, πώς θα προστατεύουμε τα δεδομένα χωρίς προστατευτισμό. Άντωνη, από εκεί που μείναμε πριν. Θα απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις ε, και ε, θα αναφερθώ και σε κάποια θέματα που είπε και ο Ανδρέα. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να συζητήσω που έκανε το παραλυσμό ανάμεσα στην αστρολογία και στην αστρονομία. Ε, ας απαντήσω στο ερώτημα της Αντιπροέδρου Μαγκίνες. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ καλή ερώτηση, διότι έχουμε συνηθίσει να ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι νομοθέτες ε, υφίστανται lobbying από πολλούς. Πολλές ομάδες ε, συμφερόντων προσφεύγουν σε αυτούς και τους πιέζουν. βρισκόμαστε σε θέση όπου έχουμε δει άνευ προηγουμένου αλλαγές. Κάποιοι παράγοντες έχουν αναπτύξει ε, ε, ε, προϊόντα, αγαθά παγκόσμια στον καράζ τους στην Καλιφόρνια. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ε, μπορούμε να ευχόμαστε να μην είχε συμβεί αυτό. Ε, σίγουρα όχι αν κάποιος είχε τον καράζ ε, και τώρα φέρει στους στους ώμους του το βάρος όλου του κόσμου και δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Επίσης αυτό ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν κάποιος νομοθετεί, ε, όταν για παράδειγμα είναι κανείς ευρωβουλευτής εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο με τις ευθύνε που έχετε. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Εγώ θα ισχυριζόμουν ότι σημαίνει ότι όσοι συμμετέχουν στον ιδιωτικό τομέα ε, συμμετέχουν σε έναν κόσμο διαφορετικό από ό,τι παλιά. Πράγματι φέρουν στους ώμους τους το βάρος των ανησυχιών όλου του κόσμου. Και όταν λαμβάνει κανείς υπόψη τα όσα γίνονται στην ε, επιχειρηματική κοινότητα, ε, στρογγύλη τράπεζα επιχειρήσεων, τι ενδιαφέρει και τις δύο πλευρές. Εάν βρίσκεστε στη θέση όπου ε, έχετε στους ώμους σας τις ανησυχίες όλου του κόσμου, βρίσκεστε στη μία πλευρά, την ιδιωτική ας πούμε, ε, ή από την άλλη υπάρχει εδώ και μια σύγκληση συμφερόντων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν νομοθετικές ομάδες στις μεγάλες παγκόσμιες πλατφόρμες. Ε, δεν ε, έχω εντρυφήσει πολύ στο θέμα αυτό. Ίσως ο Αντρέα ξέρει περισσότερα, ίσως εσείς ξέρετε περισσότερα. Δεν μιλάμε όμως για λόμπι. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που ανοίγουν γραφείο εδώ στι Βρυξέλλε ή στη Washington, ε, σας επισκέπτονται. Είναι άνθρωποι που προσπαθούν να καταλάβουν την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που συζητάμε εδώ. Έχουν ε, τις δυνατότητες αυτές. Έχουν ε, τις δυνατότητες, υφίστανται και την πίεση όμως και μάλιστα ε, πιθανότατα αυτοί να νιώθουν περισσότερο την πίεση από ότι οι κλασικοί νομοθέτες, διότι ποιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή ε, στο στόχαστρο. Ε, εντάξει, όλοι λέγανε πάντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βιαστείτε να ρυθμίσετε τα πράγματα, να νομοθετήσετε, αλλά τώρα είναι ανάποδα τα πράγματα. Συνήθως ε, λέγανε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να φροντίσει να νομοθετήσει σωστά. Και την ηρωνία την ανέφερε και η Επίτροπος Βέσταγκερ. Οι επιχειρήσεις οι ίδιες ζητάνε ρύθμιση και νομοθεσία με τρόπο άνευ προηγουμένου. Και αυτό εμένα με κάνει να σκέφτομαι ότι έχουμε έναν φυσικό σύμμαχο εδώ, μια φυσική συμμαχία ανάμεσα σε όσους θέλουν να γίνει σωστή νομοθεσία. Δεν είμαι αφελής, αλλά μιλάω για τους πραγματικά μεγάλους παράγοντες. Ε, πολλά διακυβεύονται. Δεν νομίζω ότι τους ε, συμφέρει να γίνει λάθος η νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι η φήμη τους ε, θα επιβίωνε εάν γίνονταν λάθος τα πράγματα. Το διακύβευμα είναι υπερβολικά υψηλό. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σε πολύ περίεργη θέση. Πρέπει να ε, υπάρξει επανευθυγράμμιση. Τι σημαίνει αυτό για εσά ως νομοθέτες όταν σας προσεγγίζουν αυτές οι πλατφόρμες. Αντρέα, διάβασα το βιογραφικό σου νωρίτερα ε, που ε, έχει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Google. οι ενδιαφερόμενοι, οι συμφεροντούχοι δεν έχουν πολλές επιλογές. Νομίζω λοιπόν ότι έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις. Ε, είναι και θέμα πόρων ε, και άκουσα τον κύριο Έιλερ να αναφέρει το θέμα αυτό. Μιλήσατε για τους οικονομικούς πόρους, ε, τους διαθέσιμους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να μην είναι τελείως ε, ασήμαντη, βέβαια μπορεί να μην είναι και ό,τι θα επιθυμούσε κανείς, αλλά τι ε, πόροι υπάρχουν που θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν προς όφελος του κοινού. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά με τρόπο ανοιχτό, χωρίς προκαταλήψεις χωρίς να θεωρήσουμε ότι όλα αυτά θα είναι για ε, κακούς σκοπούς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ε, ε διαθέσει κανείς τους πόρους ε, με τρόπο ώστε να αποφύγει κανείς τη σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να περίμενε κανείς. Ε, αυτή λοιπόν είναι η πολύ ενδιαφέρουσα θέση στην οποία βρισκόμαστε. Δεν βρισκόμαστε, δεν έχουμε ξαναβρεθεί στη θέση αυτή. Σίγουρα θα ε, απαιτήσει αυτό να σκεφτούμε με ανοιχτό τρόπο. Ε, έχουμε πολλές επαφές με ε, τους παράγοντες αυτούς. Ε, ε στον ΟΣΑ τους βλέπουμε παντού. Θεωρούν ότι ο ΟΣΑ αποτελεί σημαντικό στοιχείο της λύσης. Γιατί, δεν το λέω αυτό επειδή δουλεύω στον ΟΣΑ. Τι προσφέρει ο ΟΣΑ που δεν μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΟΣΑ είναι παγκόσμιος οργανισμός. Και η Εύα είπε ότι χρειαζόμαστε παγκόσμια πρότυπα. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύξει πρότυπα, δεν μπορεί να θεωρήσει ότι είναι από μόνο του παγκόσμια. Δεν είναι. Θα είναι πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ λογικό. Και άλλωστε, αν καταφέρετε να πετύχετε πρότυπα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση ε, μπράβο. Αλλά α το δούμε διαφορετικά. Ας υποθέσουμε ότι ε, έχουμε κάποιο, κάποια περιφέρεια του κόσμου που ηγείται όσον αφορά την δημιουργία προτύπων. Ε, έχει περισσότερη πείρα, έχει περισσότερους φορείς, έχει περισσότερες διαδικασίες. Και φυσικά μιλώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολείται με το παιχνίδι αυτό ε, πάνω από 50 χρόνια. Έχουμε λοιπόν ένα μοναδικό παράδειγμα. Έχω εργαστεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω αναπτύξει πρότυπα. Είχα όμως ε, και επαφές με το υπόλοιπο του κόσμου, πώς μπορούμε λοιπόν ε, να ε, συμφιλιώσουμε τις διαφορές, να χειριστούμε τις αντιθέσεις. Το... Αυτό που αλλάζει λοιπόν τώρα πια είναι ο κανονισμός προστασίας δεδομένων. Η πρώτη φορά βλέπουμε ένα πρότυπο Ε, είναι, ε, που μάλιστα ε, έχει ένα σωρό μειονεκτήματα. Είναι ένα ακρονίμιο που κανείς δεν καταλαβαίνει. Στις Βρυξέλλες έχει εκπονηθεί Υπάρχουν ε, άνθρωποι που αποχωρούν ε, σήμερα από το κτίριο για πρώτη φορά, ε, που αποχωρούν για τελευταία φορά. Όλοι αυτοί θα μπορούν να κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τι γίνεται, θα γίνει αυτό ένα παγκόσμιο πρότυπο. Και διαφωνώ με τον Ανδρέα, ίσως διαφωνώ με τον τρόπο που το είπε. Μίλησε ε, για την ε, δύναμη της ενιαίας αγοράς. Ε, αυτό δεν εμπόδισε ποτέ ούτε τους Αμερικανούς να αντισταθούν, δεν εμπόδισε εμπορικές κυρώσεις κλπ. Νομίζω ότι έχουμε το πλεονέκτημα της σωστής στιγμής του σωστού χρονοδιαγράμματος ε, και το να έχουμε ε, κάτι το οποίο όλοι χρειάζονται ε, που δεν έχουν χρόνο όμως να το εκπονήσουν. Οι Αμερικανοί δεν έχουν χρόνο για κάτι τέτοιο ξαφνικά, ούτε άλλοι. Λένε λοιπόν ότι η δημόσια πίεση επάνω μας είναι τεράστια. Ας το αρπάξουμε λοιπόν. Εάν 28 χώρες συμφώνησαν, δεν μπορεί να είναι και τόσο κακό. Ας το σκεφτούμε. Και ας κάνουμε από εδώ παρεκβολή, να κρατήσουμε το στοιχείο όπου ε, έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο μπορεί να μην ε, ε, το έχουμε και στην τεχνολογία, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως μοχλό και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά σε βάθος χρόνου. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάτι που αποτέλεσε πρωτοπορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να εξυπηρετήσει παγκόσμιους σκοπούς. Ε, έτσι λοιπόν μπορεί ο Ωσά να είναι πάρα πολύ χρήσιμος διότι ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Οι Ιαπωνέζοι μας εμπιστεύονται, οι Κορεανοί μας εμπιστεύονται, οι Κορεάτες, ε, η ε, Νέα Ζηλανδία, η Αμερική μας εμπιστεύεται, οι Καναδοί, οι Μεξικανοί, οι Χιλιανοί, οι Ισραηλινοί ε, και θα μπορούσα να συνεχίσω να απαριθμώ όσους μας εμπιστεύονται. Ακόμη και εδώ. Έχουμε 22 από τα 37 κράτη-μέλη του ΩΣΑ ασχολούμαστε με τον ψηφιακό φόρο. 140 χώρες συνεργάζονται μαζί μας ε, για να αποφύγουμε ε, έναν ε, παγκόσμιο φορολογικό πόλεμο, να έχουμε ειρήνη και να μπορέσουμε να έχουμε τα φορολογικά έσοδα που θα διευκολύνουν τον κύριο Έλερ που έχει πολύ λίγα, λίγους πόρους για παράδειγμα για την κβαντική μηχανική και όλα τα άλλα πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Υπάρχει λοιπόν χώρος και για τη την δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε εδώ τον ΣΤΟΑ, έχω ε, συμμετάσχει σε πολλές ε, συνεδριάσεις. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα καλά στοιχεία, αυτά που έχουν γίνει καλά, που αντικατοπτρίζουν τις αρχές μας, που βρίσκονται πολύ κοντά στις αρχές που αναπτύχθηκαν από την ομάδα όπου συμμετείχε ο Ανδρέα. Ε, τις ε, διαφορές αυτές ε, μπορούμε να τις επιλύσουμε και να συμφωνήσει και οι Ηνωμένε Πολιτείε που είναι μέλος του ΟΣΑ, ο Καναδάς, η Κίνα μετά. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας μεταφέρω αυτές ε, τις σκέψεις, αυτούς τους προβληματισμούς, ε, διότι έχει να κάνει με το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει το ρόλο της. Μην πέσετε όμως στην παγίδα απλά να κοιτάτε τους εαυτούς σας συνέχεια, διότι όλα αυτά θα εξυπηρετήσουν ένα υψηλότερο καλό κάποια στιγμή, εκτός... αν θέλετε να συνεχίσετε να έχουμε κατακαιρματισμένη βαλκανοποιημένη κατάσταση. The interpretation can stop. Thank you. Θα σταματήσει η διερμηνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσετε παραμένο, παραπάνω χρόνο. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. The standards and the way you put it to serve a global purpose could actually be the key to success, uh, successful setting of global standards. Um, I don't know if you would like to have